be adopted. Uh, number two, Chairman's announcements, uh, Brexit. Uh, the vote is postponed to the first or... Η ψηφοφορία αναβάλλεται για την 1η 2η Απριλίου. Και, και να δούμε γιατί πρέπει να ψηφίσει και το Βρετανικό Κοινοβούλιο και θα δούμε αν θα γίνει αυτό. Μετά περνάμε στις εκτιμήσεις ε, εσόδων και δαπανών για το 2020. Ε, ο κύριος Μάνκα είναι ο εισηγητής και ευχαριστούμε πολύ Βλάντιμιρ. Είχαμε μια πολύ δύσκολη συζήτηση με το Προεδρείο και νομίζω ότι συνολικά μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Λοιπόν, ξεκινάω αμέσως με την ψηφοφορία εάν συμφωνείτε ή όχι. Ξεκινάμε λοιπόν με μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στις πραγματικές ψηφοφορίες. Παράρτημα 1. Η θέση του εισηγητή είναι συν. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογίες του εισηγητή που περιέχουν και τη συμφωνία με το Προεδρείο με μία ψηφοφορία. Παράρτημα 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία των τροπολογιών. Ξεκινάμε. Παρά με την τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Παραγραφός 4, τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτονται. τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτονται. τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την επαληθεύσουμε. Ναι, πρέπει να τελειώσει η ψηφοφορία. Έχετε φέρει κάρτα. Όχι. Πέρας. Κατά. Οπότε είναι ισοψηφία, οπότε απορρίπτονται. Τριάντα Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε πέρας εγκρίνεται 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές να την επαληθεύσουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Είκοσι ένα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά Αποχές. Να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. «34, 35 και 36». Α, όχι. Μόνο οι 34 και 35. Ναι, πέρας. Εγκρίνεται. Με 36 καταπίπτει. 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτεται, 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την επαληθεύσουμε. Πέρας. εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 47. 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 45. Με προφορική τροπολογία του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε άρχεται πέρας εγκρίνεται 49 αποσύρεται 50 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με μια ψήφο διαφορά. Όχι. Α, απορρίπτεται. Μάλιστα. Ο κύριος Κάρας. Ωραία. 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία Μάλιστα. Ε, πίπτη μου λένε εδώ, γιατί έχει εγκριθεί η 58. Οπότε περνάμε στην 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να την επαληθεύσουμε, εντάξει. Πέρασε. Απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παραγράφος 23. Προφορική τροπολογία του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την επαληθεύσουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66 καταπίπτει. 67 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 68. Θέλετε έλεγχο, μάλιστα. Την 67. Την ελέγχουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά. Εποχές. απορρίπτεται. 69 υπέρ κατά εποχές να ελέγξουμε. Λήξη. Απορρίπτεται. 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 71, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 3, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 85. Υπέρ. Με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 85. Λήξη. Εγκρίνεται. 87 υπέρ. Καταπίπτει. 83. Υπέρ. Okay. Yes, next one. Next one. Yes. Ματική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε στο δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στην 86 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε την 99. Απορρίπτεται. Σαφέστατα πάμε στην 89 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 90. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 91 υπέρ. Με την προφορική τροπολογία κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 96. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 95 καταπίπτει. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Για την 97. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 101. Με προφορική τροπολογία από τον εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 103. Ψηφορία σε τμήματα και πάλι. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Πρώτο τμήμα για την 103. Λήξη. Εγκρίνεται. Μάλιστα, ευχαριστώ. Τότε περνάμε στο δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Καταπίπτει. Περνάμε στην 104 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 104. Άρχεται η ψηφοφορία. Κάποιος λείπει, ένας λείπει. Λήξη. Απορρίπτεται. Πάμε στην 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε στις ατυλογικές σκέψεις. 1 υπέρ. Κατά. Ανάποδα τα είπε ο Πρόεδρος. Ποιος είναι κατά, ποιος είναι υπέρ. Για να το κάνουμε αντίστροφα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Δύο λείπουν. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Όχι, εγκρίνεται. Τρία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία, με ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ, άρχεται ψηφοφορία. Ωραία, λήξη. Συγχαρητήρια στον κύριο Μανικά. Εγκρίνεται. Περάσουμε στο σημείο 4. Πρώτος κανονισμού του Συμβουλίου για την ε, λήψη κέντρου σχετικά με την κλασική και την προπολογισμό τη Ένωση σχέση με την υποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου αναβάλλεται πιθανότατα για την 1η ή τη 2η Απριλίου. Περνάμε στον προπολογισμό τμήμα 3 με τον κύριο Βιώτη, ο οποίο απουσιάζει σήμερα. είναι γενικός εισηγητή για το προπολογισμό, αν συμφωνεί ο γενικός εισηγητή, Παρακαλώ, η Έντε θέλει κάτι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, πολύ γρήγορα. Έχουμε δύο αιτήσει μεταφορά στην υπαριθμόν 5 που μεταφέρει 5 εκατομμύρια στο μέσο, από το μέσο εταιρική σχέση στο μέσο αναπτυξιακή συνεργασία για να ε, έχουμε την εμπορική συμφωνία με την Αφρική και το δεύτερο είναι μια μεταφορά που συζητήσαμε την περασμένη εβδομάδα. Θέσαμε διάφορες ερωτήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει να κάνει με 370 εκατομμύρια σε αναλήψει υποχρεώσεων για τη χρηματοδότηση δράσεων στο άσυλο και τη μετανάστευση και είχαν μείνει εκρεμείς, ε, όμως την περασμένη φορά και γραπτό και προφορικά απαντήθηκαν ερωτήσεις και ο εισηγητή μα είπε ότι ήταν ικανοποιητικέ οι απαντήσει. έτσι λοιπόν η πρότασή του είναι να υπερψηφίσουμε και τις δύο αυτές αιτήσει μεταφοράς. So I will open the vote. Ωραία, ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ, παρακαλώ. Α, ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε για την ονομαστική ψηφοφορία και για τα δύο, μια και έξω όμως. Ψηφίστε παρακαλώ. Άλλοι δύο πρέπει να ψηφίσουν ακόμα. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Και τα δύο κονδύλια. Συγχαρητήρια στον κύριο Βιώτη. Και πάμε στο επόμενο θέμα. Εγώ είμαι εισηγητή. οπότε γίνομαι εισηγητή τώρα. Και εδω έχουμε μία μεταφορά C1. Ε, το συζητήσαμε στο τελευταίο Προεδρείο και περιλαμβάνεται στο 2020, πρόκειται για 51 θέσεις για 4 εκατομμύρια και κάτι. Νομίζω το πρώτο είναι του Κοινοβουλίου, είναι γραμμή 1632, κοινωνικές ε, σχέσεις και κοινωνικές ε, δραστηριότητες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει για το 2019 και το τρίτο είναι για την ε, Ombudsman που είναι αλλαγή στις θέσεις Πρόκειται από το 86 ε, μη μόνιμος διοικητικός. Εγώ είμαι υπέρ και των ε, τριών ετοιμάτων. Πρώτα για το ΣΥΕΝΑ πρέπει να ψηφίσουμε. Ψηφίστε παρακαλώ με ονομαστική ψηφοφορία. Κατά. Α, όχι. Είναι ηλεκτρονική είπαμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Λείπουν κάποιοι. Ψηφίστε. Τέλος. Ωραία, εγκρίθηκε. Τώρα ποιο έχει αντίρρηση για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή Ομπούτσμαν. Όχι, οπότε εγκρίνεται. Και έτσι ολοκληρώνουμε. Η κυρία Χλουμάγερ δεν είναι εδώ και δεν έχει στείλει τίποτα. Είναι εδώ ο κυρία Χολμαγερ. Α, Μόνικα, μπράβο, πάνω στην ώρα. Δεχόμαστε ό,τι ήθελες. 2 Απριλίου είναι η επόμενη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.